Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας με μια μικρή καθυστέρηση. Έχουμε πολλά σημεία, πολλά ποιοτικά σημεία στην ημερήσια διάταξη. Σήμερα το πρωί έχουμε μαζί μας τον Μάτζεφ Ποπόφσκι, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Μαζί του λοιπόν θα συζητήσουμε Καταρχάς, τις τελευταίες εξελίξεις της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά το επιχειρησιακό της κομμάτι, και στη συνέχεια παρουσία του θα συζητήσουμε την ετήσια έκθεση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας. Στη συνέχεια θα συνεδριάσουμε με τους συναδέλφους μας από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Κλεισμένων των Θυρών, παρουσία της Λέδης Άστον, της ΣΥΠΑ, της εκπροσώπου για την πολιτική ασφάλεια και τις ε, εξωτερικές ε, σχέσεις και σήμερα το απόγευμα θα έχουμε την ε, κυρία Κλοντ Φρανσαρνού, εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας, καθώς επίσης και τον κύριο Χούμπρεκτ, αναπληρωτή διευθυντή του Κοινού Οργανισμού Συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών. Αύριο θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τις δύο εκθέσεις της υποπιτροπής μας, του κυρίου Κέλλαμ όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και του κυρίου Τάραντ όσον αφορά τις ε, κλιματικές αλλαγές και την ε, κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Αν δεν υπάρχουν ε, άλλα σημεία τα οποία θέλετε να προσθέσετε, ξεκινάμε υποδεχόμενοι τον κύριο Ποπόφσκι, με τον οποίο έχουμε συχνές επαφές όσον αφορά την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε ιδιαίτερα στην περιοχή του Σαχέλ, κυρίως στο Μαλί, αλλά επίσης να βερθούμε και στο ζήτημα της Συρίας είναι τα δύο βασικά ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα και θα μπορούσαμε επίσης να αναφερθούμε και στις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας, κυρίως στο Κέρα, της Αφρικής και στο Σαχέλ. Έχουμε μια νέα αποστολή στην Νιγηρία, στον Νίγηρα με συγχωρείτε, και θα μπορούσαμε επίσης να έχουμε και μία αποτίμηση της συνεδρίασης των Υπουργών Άμυνας που έγινε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Θα αναφερθούμε έπειτα στη συνέχεια, όπως σας είπα, και στην ετήσια έκθεση. Κύριε Ποπόφσκι, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα αλλάξω λίγο τη σειρά της παρουσίασης. Θα κάνω την ενημέρωση για την Υπουργική Διάσκεψη στην αρχή και μετά θα επικεντρωθώ σε διάφορα σημεία και εδώ είμαι και με τον συνάδελφο ο οποίος είναι ε, Γενικός Διευθυντής ε, του IMS και με το Hansel Κάβελ του ECCC. Επομένως, αν υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και κάποιες ε, λεπτομέρειες. Ξεκινώντας λοιπόν με την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έγινε στην Κύπρο στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στην ημερήσια διάταξη είχαμε τρεις ε, συνεδριάσεις, ε, μία που αφορούσε την ε, νότια γειτονία, αλλά με πολύ ευρύς όρους, γιατί συζητήσαμε για την περιοχή και μετά την περιφερειακή διάσταση και τις δυνατότητές μας. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη ε, επικεντρώθηκε κυρίως στη συζήτηση ε, στο Σαχέλ και στο Μαλί. Ήδη από τότε, στην ημερομηνία της συνεδρίασης, διαπιστώνουμε ότι υπήρχε, αν όχι η συνένεση, η κατάλληλη στιγμή για να ληφθούν αποφάσεις ε, για δέσμευση πρωτίστως. Οι Υπουργοί συζητούσαν το θέμα της στήριξής μας στην ΕΚΟΓΟΣ την οικονομική κοινότητα των δυτικοαφρικανικών χωρών και τη σταθερότητα στην περιοχή και τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, ανοικοδόμηση και την ε, ε, αναδιάρθρωση του στρατού του Μαλή. Όπως ξέρετε, μας προσέγγισε και η ΕΚΟΓΟΣ και ζήτησε στήριξη ένα, αλλά με πολύ ευρύς ακόμα. Πρέπει λίγο να δούμε τις λεπτομέρειες. Και αμέσως πριν την Υπουργική Διάσκεψη, ο υπηρεσιακός πρόεδρος και πρωθυπουργός του Μαλή απέστειλαν έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας ε, πολύ συγκεκριμένη συνδρομή και σε θέματα επιμελητίας ε, και χρηματοοικονομική και υλική στήριξη ε, για το στρατό στο Μαλή. Αυτά λοιπόν ήταν τα θέματα υποσυζήτησης. Σε γενικές γραμμές οι Υπουργοί Άμυνα συμφώνησαν να εξετάσουν τις εναλλακτικέ τους λύσεις. Ε, υπήρχαν αρκετές ε, ε, θέσεις. Πολλοί θεώρησαν ότι ναι, μένει είναι κατεπήγον, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν δομές για να μπορέσει να συμμετάσχει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση με βοήθεια. Υπάρχει όμως και το σχετικό ψήφισμα ε, στον ΟΗΕ. Υπάρχει ένα σχέδιο ψηφίσματος το οποίο πρόκειται να συζητηθεί κατά πάσα πιθανότητα σήμερα. Αυτά είναι τα τελευταία νέα που είχα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σύντομα μπορεί να έχουμε ψήφισμα. Α, δεν έχει όμως επιβεβαιωθεί ακόμα. Αυτή είναι η πρώτη παράμετρος. Και από εκεί και πέρα υπήρχε και το δεύτερο στοιχείο που είναι η τοπική αφρικανική ιδιοκτησία. Θα πρέπει ε, να υπάρχει εντολή για την αποστολή. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη. Έγιναν κάποιες προκατακτικές συζητήσεις και κατόπιν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο την επόμενη εβδομάδα στις 15 Οκτωβρίου δεν έχουν ακόμα ληφθεί αποφάσεις, αλλά ένα από τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί επιτάπητος ε, είναι ότι μπορεί να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, να αναπτύξει ε, μία δομή αντιμετώπισης κρίσεως από το Συμβούλιο ε, Εξωτερικών Υποθέσεων που θα γίνει τον Νοέμβριο. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που συζητήσαμε. Και οι Υπουργοί κατέληξαν ότι θέλουν να έχουν ε, ε, ένα πλήρες μενού εναλλακτικών λύσεων. Έτσι το αποκάλεσε ο Γάλλος υπουργό. Θέλουμε να εξετάσουμε λοιπόν το θέμα της χρηματοοικονομικής στήριξης στην ΕΚΟΓΑΣ. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε λίγα περισσότερα πράγματα για αυτήν. Και επίσης ε, εκπαίδευση του στρατού στο Μαλί. Υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο είναι πολύ γνωστό. Είναι η αποστολή εκπαίδευση του στρατού του EUTM. Έχει ε, ε, ξεκινήσει, είναι να εξελίξει ε, στην Ουγγάντα για αρκετό καιρό για πρώην ε, στρατιωτικούς του Μαλή. Ε, πρέπει βέβαια κάπως να προσαρμοστεί κάπως και θα πρέπει να καθοριστεί και σαφώς τι εντολή θα έχουν. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν πρέπει να υπάρχει και δέσμευση από πλευράς αρχών ε, στο Μαλή. Θέλουμε επίσης να το θέσουμε και στο ευρύτερο πλαίσιο της γενικότερης κατάστασης στο Μαλή ό,τι και να κάνουμε ε, από πλευράς επιχειρησιακής δέσμευσης θα πρέπει να είναι τμήμα ενός χάρτη πορείας προς τη σταθερότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι σαφές ε, για όλα τα κράτη-μέλη. Θα θέλαμε ο χάρτης πορείας να οδηγήσει σε εκλογές στο Μαλί και από εκεί και πέρα η κυβέρνηση στο Μαλί θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα ήθελε να σταθεροποιήσει την κατάσταση και στο Νότο, αλλά ιδίως ε, στο βορρά της χώρας. Και εμείς φυσικά θα είμαστε στη διάθεσή τους για να τους ε, βοηθήσουμε. Η συζήτηση λοιπόν ε, σίγουρα θα συνεχιστεί την επόμενη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο. Τώρα, για τη Συρία δεν υπήρχαν και τόσο πολλά θέματα προς συζήτηση οι Υπουργοί αναφέρθηκαν ε, στο κίνδυνο διάδοσης και χρήσης χημικών όπλων. Η κατάσταση εξακολουθεί να επιδεινώνεται και γνωρίζουμε φυσικά ότι η Συρία έχει αποθεματικό χημικών όπλων, τα οποία είναι έτοιμα προς χρήση, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ε, σχέδιο αντιμετώπισης μιας τέτοιας κατάστασης. Παρακολουθούμε όμως πάρα πολύ στενά την κατάσταση. η κατάσταση στο Νότο που συζητήθηκε και συζητάται ακόμα στο Συμβούλιο είναι ε, η κατάσταση της Λιβύης. Ε, βέβαια το θέμα διονύζεται, το γνωρίζουμε. Έχουμε ήδη ε, αναπτύξει μία αποστολή ειδικών των εξωτερικών συνόρων. Αυτό ήταν τμήμα της προσπάθειας των Ηνωμένων Εθνών και των χωρών της Λατινικής Αμερικής και ε, προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε ένα θέμα αντιμετώπισης ε, κρίσεων για τη διαχείριση των συνόρων και την ασφάλεια στη Λιβύη. Θα πρέπει βέβαια να υπερβούμε και κάποιες δυσκολίες ε, όσον αφορά την διεξαγωγή μιας ε, αποστολής για να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει επί τόπου. Ε, έχουμε ειδικού οι οποίοι είναι έτοιμοι ε, να πάνε, αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ ρευστή η πολιτική κατάσταση στη Λιβύη. Περιμένουμε να σταθεί νέα κυβέρνηση η οποία θα συνεργαστεί μαζί μας και θα συμφωνήσει επί των παραμέτρων της συνεργασίας. Ξέρετε όμως ότι ο νέος ε, πρωθυπουργός δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση και χρειάστηκε να παραιτηθεί. Αυτό νομίζω έγινε χθε. Υπάρχει λοιπόν πολιτικό κενό και είναι πολύ δύσκολο να ε, μεταβούμε διότι δεν υπάρχουν συνομιλητές και μια αντίστοιχη κατάσταση αντιμετωπίσαμε και την Άνοιξη. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη λοιπόν τα οποία ανυπομονούν και δε ότι πρέπει να δράσουμε, αλλά από την άλλη πρέπει να υπάρχει και συμμετοχή από πλευράς ε, Λιβύης. Ε, και η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη. Παρακολουθούμε βέβαια πολύ στενά την κατάσταση με την αντιπροσωπεία μας στην Τρίπολη, η οποία παρεπιπτόντως ενισχύθηκε με δύο ειδικού ασφαλείες οι οποίοι είναι ήδη επιτόπου και εξετάζουν ε, τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και τη διαχείριση των συνόρων. Ε, μπορούν να κάνουν ελάχιστα βέβαια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά αυτό τη συνήθη διαδικασία προετοιμασίας ε, για μια αποστολή του CSTP τη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Τώρα, για τι υπόλοιπε αποστηλίε, το κέρα τη Αφρική. Εκεί ήταν λίγο καθησυχαστικά τα πράγματα για μας. Ε, ακούσαμε ότι τα κράτη-μέλη είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιημένα με την πρόοδο και τις δράσεις που γίνονται για τις αποστολές και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ε, επιτόπου. Και αυτό το Ακούσαμε και με, από τους επικεφαλείς της αποστολής ε, ε Αταλάντα και από τον επικεφαλής της EU Καπνέστορ που είναι ο νέος ε, υπεύθυνο ε, της αποστολής που μόλις ξεκινάει αλλά θέλουμε να έχουμε και στοιχεία και από αυτόν. Αναγνωρίστηκε λοιπόν ότι έχουν υπάρξει επιτεύγματα από πλευράς μας αλλά γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει ε, περιθώριο να είμαστε πιο συγκαταβατικοί για τα θέματα της πειρατείας, επομένως πρέπει να συνεχιστεί η αποστολή. Η Αταλάντα θα συνεχίσει για δύο ακόμα χρόνια. Ε, η αποστολή UTM ήταν αρκετά επιτυχή στη Σομαλία και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους και στο τέλος της ε, εντολής αυτής θα έχουμε εκπαιδεύσει αρκετές χιλιάδες Σομαλούς στρατιώτες και Κάποιοι από αυτούς βρίσκονται ήδη και συνεργάζονται με τα στρατεύματα της, ε, ε, που βρίσκονται εκεί. Υπάρχει αρκετή πρόοδο στις τελευταίες εβδομάδες, αλλά φυσικά έχουμε και αρκετά ακόμα πράγματα να κάνουμε και κάτι το οποίο προέκυψε, το οποίο πρέπει να εξετάσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια όταν θα γίνει η αναθεώρηση της αποστολή και θα επανέλθουμε στα κράτη-μέλη για το κατά πόσον θα πρέπει να παραταθεί η αποστολή κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αλλά πρέπει να αποφασιστεί, ε, είναι το γεγονός ότι κάποια κράτη-μέλη θεωρούν ότι τμήμα της προσπάθειας της εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνεται στη Σομαλία, στο Μογκαντούισου. Ε, χρηματοδοτήθηκε ε, και ένας χώρος ε, ε, για, τις, ε, για την εκπαίδευση στο Μογκαντήσου, το στρατόπεδο Τζαζίρα, το οποίο λογικά θα είναι έτοιμο. Αλλά αυτό είναι το μήνυμα το οποίο προέκυψε από αρκετέ χώρε μέλη. Χρειάζεται βέβαια να έχουμε και μια πολύ καλή ανάλυση κινδύνου για οποιαδήποτε μεταφορά δραστηριοτήτων στη Σομαλία πριν ληφθεί απόφαση. Αυτό βέβαια θα πρέπει να το μελετήσουμε στις επόμενες 4 με 5 εβδομάδες, διότι πρέπει να ληφθεί απόφαση ε, και τέλος, οι υπουργοί ε, συζήτησαν και την αποστολή Αλθέα. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο, διότι πρέπει κάθε φορά να ε, συζητάμε και με τα Ηνωμένα Έθνη για απόφαση για παράταση της εντολής και κάθε φορά αυτό το οποίο προκύπτει είναι κατά πόσον θα πρέπει να παραμείνει η εκτελεστική εντολή ε, της αποστολής. Ε, η Αλθέα βέβαια έχει υποβαθμιστεί και η διαδικασία έχει αναδιαμορφωθεί και πλέον ε, έχει υλοποιηθεί η νέα αναδιαμόρφωση. Ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Έχουμε πλέον 600 στρατιώτες, αλλά αυτό το οποίο οδήγησε την ύπατη εκπρόσωπο να προτείνει να παραμείνει η εκτελεστική εντολή για ένα ακόμα χρόνο ήταν ε, το πολιτικό πλαίσιο για την κατάσταση στη Βοσνία είναι ακόμα σταθή. Και η αποστολή είναι σταθεροποιητικός παράγοντας για πολλούς λόγους ε, πολιτικής φύσεως και αυτό το οποίο ε, κατέστη σαφές είναι ότι από στρατιωτικές πλευράς τα πράγματα είναι σταθερά. Αλλά θεωρείται απαραίτητη η παρουσία. Τα κράτη-μέλη βέβαια είναι διαιρεμένα, υπάρχει διάσταση απόψεων ε, ως προς τις ε, χονδρικές ε, γραμμές που πρέπει να τηρηθούν, αλλά πιστεύω ότι θα υπάρξει συνένεση πριν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, το θέμα των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Υπήρχε συζήτηση για το pooling and sharing, θα ακούσετε πολύ περισσότερα από τον Κλοντ Φλανσουάρνο σήμερα το απόγευμα, αλλά η υπηρεσία επί τη ευκαιρία της συνεδρίασης πρέπει να γίνει μια συζήτηση για ένα κώδικα διοντολογίας για το pooling, sharing, pooling and sharing, ένα βασικό κώδικα διοντολογίας. Δεν είναι ληφθή απόφαση γι' αυτό, είναι πολύ νωρί, αλλά η βασική αντίδραση των κρατών μελών ήταν θετική, αρκετά θετική. Και ε, Ελπίζω το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού να συμφωνήσει για αυτό τον κώδικα τον Νοέμβριο. Η φέρπουσα υπόθεση είναι ότι το pooling and sharing θα πρέπει να είναι τμήμα του, ε, της διαδικασίας του εθνικού σχεδιασμού άμυνας. Ε, δεν είναι κάτι καινοφανές. Ε, η EDA ασχολείται με το θέμα αυτό και προσπαθεί να το επιτύχει τα τελευταία 15 χρόνια ε, και υπήρχε και μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση από τη Σουηδία γιατί νομίζω ότι είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ήδη κάνει αυτό τον επίσημο σύνδεσμο. Η διαδικασία άμυνας της Σουηδίας, το εθνικό της σχέδιο, περιλαμβάνει και τον, τον εξορθολογισμό του pooling and sharing και το ίδιο θα θέλαμε να κάνουμε και τα κράτη-μέλη. Η γενική εικόνα όμως ήταν πολύ ενθαρρυντική. Και πάλι λοιπόν για τις δυνατότητές μας, ένα ε, άλλο θέμα ε, το οποίο επανακύπτει συνεχώς είναι οι αίθουσες επιχειρήσεως οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα ε, ξέρετε ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι γι' αυτό συμπεριλαμβάνεται και χρηματοδότηση αλλά τα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα πλέον να εξετάσουν κάποιες βελτιώσεις χωρίς όμως να αλλάξει το σκεπτικό κατά πάσα πιθανότητα ε, θα συμφωνήσουν και προς τα... τη συνέχεια του έτους με την έννοια ενός ε, ε, έθνους το οποίο θα ε, παρέχει το βασικό πυρήνα της στρατιωτικής δύναμης και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι θα είναι λίγο στα μετόπιστα. Είναι αυτό βέβαια πρέπει να το εξετάσουμε ακόμα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι, να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία μιας στρατιωτικής ομάδας και όχι όλη ας πούμε την ομάδα, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό θα μπορούσαμε ίσως να χρησιμοποιήσουμε τμήματα επι, επιμελητίας, ε, ομάδα ιατρικής υποστήριξης, ε, ε, να μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τμήματα μιας στρατιωτικής μονάδας μεμονωμένα, χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε όλη τη στρατιωτική μονάδα. Όπως σας είπα δεν ελήφθη απόφαση, γιατί, αλλά ήταν πολύ χρήσιμα τα όσα ακούσαμε. Υπάρχει και συνένεση και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε κάποιες αποφάσεις ε, προς αργότερα μέσα στο έτος. Υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο μάλλον θα συζητηθεί και στη δική σας την έκθεση. Η προπτική τη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για θέματα ασφάλειας και άμυνας ε, προς τα τέλη του επομένου έτους. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Φανερόμπαϊ, σχεδιάζει να γίνει μια συνολική συζήτηση για την ασφάλεια και την άμυνα του χρόνου. Θα τα προετοιμάσουμε ήδη από τώρα και φυσικά θα πρέπει να εξετάσουμε και τι γίνεται πέραν των ε, συνήθων τμήματων που έχουμε εδώ, τις δυνατότητες εταιρικέ μας σχέσεις. Θα πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα της βιομηχανίας και των πτυχών της αγοράς, ε, να συνεχίσουμε και τα όσα έχουν γίνει μέχρι τούδε από την ε, Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Άμυνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να παρουσιάσει και μια ανακοίνωση για την αμυντική βιομηχανία κάποια στιγμή εντός του 2013 και θεωρώ ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική οπτική γωνία αν θέλουμε να έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, συζήτησε τελευταία φορά τα θέματα αυτά το 2008. Επομένως, ε, μια φορά στα πέντε χρόνια έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια συζήτηση πολιτικού προσανατολισμού σε συνολικό επίπεδο και θα ξεκινήσουμε προετοιμασία ήδη από τώρα και θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις υπορδικικές διασκέψεις από τώρα μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 για να προετοιμάσουμε το έδαφος για τη συζήτηση αυτή θα, όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να επιβεβαιωθούν και από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο ε, ε φέτος θα δώσει ειδικά καθέκοντα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας για να προετοιμάσουν τη συζήτηση αυτή για τους αρχηγούς κρατούς και, και κυβερνήσεων ώστε να μπορέσουν να τα συζητήσουν όλα αυτά το Δεκέμβριο του 2013. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ. Θα επανέλθουμε σε πολλά από αυτά τα θέματα όταν θα συζητήσουμε την έκθεση. Ευχαριστώ. Merci, merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Θα υποφεληθώ από την παρουσία του κυρίου Αμπέρ, ε, του... για να του πω ότι σε σχέση με την αποστολή στην Γεωργία, ε, η UMM ήταν στη Γεωργία στο πλαίσιο της παρατήρησης ε, των εκλογών και εκεί μας ε, είπαν πόσο θετικοί ε, αξιολογούν την αποστολή, η οποία παρόλα αυτά έλαβε χώρα σε ένα κάπως δυσχερές ε, πλαίσιο όσον αφορά τις δυσκολίες πρόσβασης στην Οσετία και στην Απχαζία ιδιαίτερως. Και ελπίζω οι εξελίξεις να μην θέσουν ένα αμφιβόλο την ε, αποστολή αυτή, το σκόπιμο χαρακτήρα της αποστολής και είναι σημαντικό να πενθυμίζουμε ε, σε τακτικά χρονικά διαστήματα να μας ε, ενημερώνουν σε σχέση με την αποστολή. Νομίζω ότι είπατε εκπρόσωπος έχει δυνατότητα να κάνει συχνά αυτή την υπενθύμηση. Τώρα, όσον αφορά τις διάφορες επιχειρήσεις, ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση όσον αφορά το κέρας της Αφρικής, όπου πράγματι θεωρώ ότι αυτά που θα κάνουμε σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο είναι πραγματικά, έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα. Ε, έχουμε αυτή την αποστολή EU Cup Nestor ε, που είναι σε περιφερειακό επίπεδο όσον αφορά τις στρατιωτικές δυνατότητες και όσον αφορά την εξέλιξη επιτόπου στην Σομαλία και την πρόοδο που έκανε η Αμισόπ η Αμισόμ όσον αφορά την σχετική σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης ε, έχει δοθεί μια προτεραιότητα στην ίδια την Σομαλία και στις δυνατότητες της ε, Σομαλίας ε, ε, είναι, μπορούμε να θέσουμε αυτό το ζήτημα ή είναι πρόημο σε αυτή τη φάση. Ε, η Πρισακίτς και ο κύριος Βάγκελ στη συνέχεια θέλουν να πάρουν το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις πλήρεις διεξοδικές πληροφορίες που μας δώσατε. Μια γενική ερώτηση θα ήθελα να θέσω. Μια γενική λοιπόν ερώτηση. Προέρχομαι από την Σουηδία. Μετά την συμφωνία για το pooling and sharing στην οποία συμμετέχει η Σουηδία, μπορούμε να χρησιμοποιούμε πλέον τους αμυντικούς μας πόρους κάτι ένα καλύτερο τρόπο και βασίζουμε επίσης και στην εμπειρία που έχουμε από τον πόλεμο στην Βοσνία. Πολλές φορές έχουμε συστήματα τα οποία επικαλύπτονται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Από τη μια λοιπόν έχουμε τη συνένωση και την κοινή χρήση, αυτή τη συνεκμετάλλευση. Από την άλλη όμως πιστεύετε ότι ε, έχουμε ήδη μια τόσο καλή συνεργασία με τον ΝΑΤΟ έτσι στο μέλλον να αποφύγουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα, να υπάρχει μια πραγματική αλληλοσυμπληρωματικότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε ένα σύστημα pooling and sharing και με τον ΝΑΤΟ έτσι ώστε σε κάποιες δυνητικές μελλοντικές διενέξεις να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει κάτι συγκεκριμένο και το ΝΑΤΟ θα κάνει κάτι άλλο, έτσι ώστε να μην έχουμε την κατάσταση που είχαμε στη Βοσνία το 1995. Τέσσερα χρόνια χρειάστηκε να περάσουν, προτού καταλάβουμε ότι κάνουμε ουσιαστικά πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Θα μπορούσε να γίνει κάτι από στη Συρία σε κάποια άλλη μελλοντική διένεξη. Ευχαριστούμε, αλλά μην ξεχνάτε ότι η CSDP δεν υπήρχε τότε. Η κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνας δεν υπήρχε. Ναι, ναι, συμφωνώ, ναι. Είναι ένα μάθημα το οποίο διδαχθήκαμε τότε. Και μετά το Κωσυφοπέδιο ουσιαστικά είδαμε ότι χρειαζόμασταν μια κοινή, πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Αυτό ήταν το τίμα το οποίο χρειάστηκε να πληρώσουμε. Ο πόλεμο στη Βοσνία ήταν το τίμα το οποίο χρειάστηκε να καταβάλουμε για να συνειδητοποιήσουμε ότι, ότι χρειαζόμαστε μια κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Ο κ. Βάγκεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω και τον κύριο Ποπόφσκι για την εκτενή του αυτή εισαγωγική παρουσίαση. Θα ήθελα να σας θέσω και εγώ με τη σειρά μου μία ερώτηση. Εμείς βασιζόμενοι στις καταστάσεις οποίες περιγράψατε στο Μαλί, στην, στο κέρας Αφρικής, στη Συρία, Μπορούμε να πούμε ότι στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας έχουμε πετύχει κάπου ένα θετικό αποτέλεσμα. Έχουμε καταφέρει να πλησιάσουμε έστω σε μία λύση, γιατί καταλαβαίνετε ότι διαφορετικά δεν την εντύπωση ότι όλοι έχουν δίκιο, ότι όλοι κάνουν αυτό το οποίο πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει, όλοι υποβάλλουν τελικά αναφορές και εκθέσεις σε εμά, στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, αλλά στην πράξη η κατάσταση εν γέννη επιδεινώνεται, βλέπουμε όλο και περισσότερες κρίσεις να ανακύπτουν. Έχουμε για παράδειγμα την ε, κατάσταση που έχει προκύψει στις σχέσεις Τουρκίας και Συρίας με τη διένεξη στην Συρία και υπάρχει μια έντονη διασύνδεση όλων αυτών των προβλημάτων. Αν δούμε το Μαλή, βλέπετε υπάρχει πίσω από το Μαλί. Ουσιαστικά η κατάσταση στο Μαλί συνδέεται άμεσα με την Δυτική Σαχάρα, Μετά τα όσα συνέβησαν στο παρελθόν στη Λιβύη. Όσον αφορά την Δυτική Σαχάρα, πήγα εκεί πέρα μία εβδομάδα μετά την εικαζόμενη αυτή απαγωγή κάποιων ανθρώπων από την Αλκάιντα. Επομένως με ενδιαφέρει πολύ το ζήτημα αυτό. Και ξέρετε ότι αναλύοντας όλα αυτά τα ζητήματα φτάνουμε και στην ισραηλο διένεξη, η οποία απλώνεται αυτή τη στιγμή όλο και περισσότερο στην Ιορδανία. Με ανησυχεί ιδιαίτερα η κατάσταση στην Ιορδανία, είμαι σε επαφή με ανθρώπους από τη χώρα αυτή η κατάσταση εκεί πέρα επιδεινώνεται και αυτό το οποίο βλέπουμε εν γέννη είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα αδιέξοδο, μη τι άλλο σε μια στασιμότητα. Ακόμα και στην ανάλυση της κατάστασης στη Συρία, όπως αυτή γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κάποιους πολιτικούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είπαν ότι θα πρέπει να βομβαρδίσουμε και ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα λύσουμε τα προβλήματα, να βομβαρδίσουμε ποιον και τι και τι αποτέλεσμα θα καταφέρουμε να αποκτήσουμε με αυτό. Νομίζω ότι μόνο ο λαϊκισμός θα μπορούσε τελικά να υποδεικνύει μια τέτοια στάση. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω πραγματικά τι γίνεται στα πλαίσια της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και τι γίνεται στο δικό σας τομέα όσον αφορά την πρόθεση να καταλήξουμε σε κάποια αποτελέσματα, γιατί αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι μόνο η μεγαλύτερη σταθερότητα και όσο δυνατόν λιγότερες διενέξεις. Αυτό θα ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν αναφερθήκατε στις ε, ευθύνε των πολιτικών. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν ποια είναι η δική σας η άποψη. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ζήμκη. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά καταρχήν ε, κύριε Υπουργέ. Ήταν πολύ σημαντικά τα όσα μας είπατε και νομίζω ότι πραγματικά άξιζε το κόπο να τα ακούσουμε όλα αυτά. Βεβαίω πάντοτε προσπαθούμε να εξετάζουμε αυτό το οποίο συμβαίνει στο χώρο της ασφαλείας, αλλά μια τέτοιου είδους συνθετική παρουσίαση είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα. Το πρώτο είναι γενικής φύσεως μάλλον και το δεύτερο είναι πιο ειδικό, έχει πιο προσωπικό χαρακτήρα. Θα ξεκινήσω με το γενικότερο θέμα. Κύριε Ποπόφσκι, εγώ δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω την άποψή σου ότι θα πρέπει να σταματήσω δεν θα πρέπει να πάψουμε να έχουμε ψευδεστήσεις όσον αφορά τις ε, μάχημες ομάδες. Ε, νομίζω ότι είναι απογοητευτικό. Ε, υπάρχουν ε, διάφορες χώρες που τις εξοπλίζουν με πραγματικά εξειδικευμένες δυνάμεις, αλλά στη συνέχεια δεν συμβαίνει απολύτως τίποτε, όλοι εφησυχάζονται, αλλά όλα αυτά κοστίζουν πολλά χρήματα και δεν επιφέρουν καμία απολύτως υπεραξία. Θα πρέπει λοιπόν ε, να, το, να αποφασίσουμε ότι είτε να τις αξιοποιήσουμε ή τελικά να τις διαλύσουμε. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε με αυτές τις ε, Δεύτερον, εγώ ήμουν κάπως ε, διστακτικός κατά πώς θα πρέπει να θέσω το θέμα αυτό εδώ στην Επιτροπή, γιατί έχει κάπως ε, προσωπικό χαρακτήρα αλλά ορισμένες φορές ε, τέτοιου είδους ε, υποκειμενικά θέματα μπορούν να δείξουν κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε κάτι ή όχι. Ε, πρόκειται για το εξή. Για το Μαλί. Αναφερθήκατε στο θέμα του Μαλί. Και εδώ, εκεί σκοτώθηκε ένας ε, νέος Πολωνός, 23 ετών, και δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο να ήταν χολέρα ή ελονοσία ε, που έφταιγε. Ε, επιτύχθηκαν ε, διάφορα σενάρια, αλλά ε, δεν ήταν δυνατόν να μεταφερθεί ισορός στην Πολωνία. Και γιατί αναφέρω το θέμα αυτό. Το Κοινοβούλιο της Επιτροπής αυτής ε, δεν είναι αρμόδιο, αλλά τέτοιου είδους περιστατικά μας δείχνουν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια υπεραξία στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ε, ας πάρουμε τα όσα είπατε κύριε Ποπόφσκι, γιατί οι βοήθειες στον τομέα της ασφάλειας και η κατάρτιση ε, μπορούν να χρησιμεύσουν και σε τέτοιου είδους ανθρωπιστικές υποθέσεις δεν μπορεί να μας βοηθήσει εδώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και σε θέματα ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Δεν πρόκειται εδώ βεβαίως για μείζωνα θέματα, αλλά καμιά φορά πραγματικά ματώνει η καρδιά μας και θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Thank you Ο κύριο Κέλα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ποπόφσκι που ήρθατε εδώ και μας είπατε τις τελευταίες πληροφορίες. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας συγχωρώ, συγχαρώ και εσάς και τις αποστολές σας που ήταν επιτυχείς ε, στο κέρας της Αφρικής και προσβλέπουμε και στη θετική μας συνεισφορά μέσω της αποστολής μας εκεί. Για τη Συρία όμως ανησυχούμε συνεχώς ε, για τις ε, συνέπειες εκεί και το γεγονός ότι η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς. Είπατε ότι δεν έχετε κάποια συγκεκριμένα σχέδια για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Ναι, μεν παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, αλλά αυτό ε, σχετίζεται μόνο στην πρόθεση για χρήση χημικών όπλων ή τη γενικότερη κατάσταση. Για τη Λιβύη τώρα, νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε την ιδέα μιας ε, πιθανής αποστολής ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας στα σύνορα. Είπατε ότι δεν έχουμε συνομιλητές αυτή τη στιγμή, αλλά θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας στην έκθεση που θα έχουμε στη συνέχεια του συναδέλφου του κυρίου Ντανζάν για τη Λιβύη, που λέει ότι στην περίπτωση της Λιβύης υπήρχε δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει με συντονισμένο τρόπο, αν χρειαστεί και σε στρατιωτικό επίπεδο, στα πλαίσια των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας αλλά δυστυχώς χάθηκε αυτή η ευκαιρία, διότι διείσταντο οι απόψεις μεταξύ των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε απλώς ρόλο παρατηρητή. Τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να υπερβούμε μια τέτοια κατάσταση. Και τέλος, για το pooling and sharing και τις μάχημες μονάδες, είπατε ότι οι Υπουργοί Άμυνας ανέφεραν την ιδέα ενός κώδικα διοντολογίας για το pooling and sharing και ε, τόνισαν ότι υπάρχει ανάγκη η όλη διαδικασία να είναι πιο συστηματική και πιο βιώσιμη όσον αφορά τα αποτελέσματα και τα ε, πρακτικά μέτρα. Ε, νομίζω ότι ακούμε συνέχεια αυτές τις καλές προθέσεις, αλλά στη συνέχεια δεν συμβαίνει τίποτα. Πόρο απέχουν από τη λύση, Υπουργοί Άμυνας. μήπως θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τι είναι αυτές οι ιδέες για πιο ευέλικτη χρήση των μάχημων μονάδων. Ε, υπάρχουν κάποια σχέδια για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των μάχημων μονάδων, όπως ανέφερε μόλις και ο συναδελφός μου. Ευχαριστώ. Yeah, Σας ευχαριστούμε. Κύριε Ποπόφσκι, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Πολλές ερωτήσεις. Θα τις απαντήσω με τη σειρά που ετέθησαν. Όσον αφορά το ζήτημα της Σομαλίας. Τα όσα σας είπα θα συμβούν στα πλαίσια της αποστολής EU Cup Nestor, η οποία θα συνεργαστεί με τις αρχές της Σομαλίας για την κατάρτιση των αστυνομικών δυνάμεων, καθώς επίσης και των κατασταλτικών δυνάμεων, των διοκτικών αρχών, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της πειρατείας. Είναι μέρος της εντολής της γενικότερης λοιπόν αυτό. Αποτελεί για μας πρόκληση να καταφέρουμε να συνεργαστούμε με χώρες οι οποίες πολλές φορές προσπαθούν να νοικοδομήσουν κάποιες βασικές δομές τους. Η αποστολή πάντως βρίσκεται στα πρώτα της στάδια και είναι ιδιαίτερα ευρία. Επομένως καταλαβαίνετε ότι η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη και αυτό ακριβώς ανέφερε και ο διοικητής της αποστολής αυτής, της επιχείρησης αυτής, να απευθύνθηκε στους Ευρωπαίους Υπουργού Άμυνα. Είπε ουσιαστικά ότι πρέπει να απευθυνθούμε σε μια πολύ μεγάλη γεωγραφική ζώνη, με πολλούς επιμέρους γεωγραφικούς κόμβους και αποτελεί ενδεχομένω την πιο δύσκολη επιχείρηση την οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε ποτέ από επιχειρησιακή τουλάχιστον πλευράς. Τώρα όσον αφορά το pooling and sharing, και την σχέση μας με το ΝΑΤΟ. Ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει πολύ συχνά και η ερώτησή σας είναι σίγουρα πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι έχουμε ήδη καταφέρει να δημιουργήσουμε έναν πολύ καλό μηχανισμό συντονισμού με το ΝΑΤΟ. Και ήδη στο παρελθόν, όταν προετοιμάζαμε εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση την σύνοδο του Σικάγο, το Μάιο, στον σύνοδο του ΝΑΤΟ, συνεργαζόμασταν σχεδόν σε καθημερινή βάση με τους εκπροσώπους του ΝΑΤΟ εδώ στις Βρυξέλλες καθώς επίσης και με τους εκπροσώπους του ΝΑΤΟ στον Όρφοκ προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να αποφύγουμε επικαλύψεις. Αν δούμε λοιπόν τα πιλωτικά προγράμματα, τους καταλόγους των πιλωτικών προγραμμάτων στα οποία καταλήξαμε, θα δείτε ότι πραγματικά έχουμε καταφέρει εκεί πέρα να πετύχουμε αυτή την ευκταία συμπληρωματικότητα. Επίση, στα πλαίσια του pooling and sharing θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι το στρατιωτικό δυναμικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε επιχείρηση και αποστολή. Όχι δηλαδή να προβλέπονται μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο για το ΝΑΤΟ. Αν υφίστανται δηλαδή ευρωπαϊκές ικανότητες και δυνατότητες, ότι θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και αντίστροφα. Αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο της κοινή αυτής συμφωνίας που έχουμε με το ΝΑΤΟ. Και αυτό το οποίο θέλουμε να προωθήσουμε την κινητικότητα, ανάπτυξη κοινών δυνάμεων και αυτό έχει συζητήσει πάρα πολλές φορές η Λέβη Άστον με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Και μιλώντας σήμερα το απόγευμα σε εκπροσώπους του ΝΑΤΟ θα αναφερθεί ακριβώς στα ζητήματα αυτά και στο pooling and sharing η ερώτηση του κυρίου Βάγγελ τώρα. Καταλαβαίνω προφανώ ότι αναφέρεστε στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό. Εξίσου όμω σημαντικό είναι να δούμε τι επιχειρήσει αυτέ και ω πλαίσιο, ω τμήμα, με συγχωρείτε, των πολιτικών μα στρατηγικών. Υπάρχει πάντα δηλαδή μια πολιτική διάσταση. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Γι' αυτό το λόγο αρχίζουμε και εργαζόμαστε στα πλαίσια ενός πολιτικού πλαισίου, όπως για παράδειγμα στο κέρας της Αφρικής. Οι εκεί αποστολές αποτελούν ένα μόνο τμήμα της ευρύτερης δέσμευσής μας. Όσον αφορά το κέρας, το κέρας της Αφρικής, είμαστε οι πιο σημαντικοί παράγοντες όσον αφορά την ανθρωπιστική συμβολή στην περιοχή αυτή. Έχουμε εκπροσώπους εκεί που συντονίζουν τις προσπάθειές μας. Έχουμε και γραφείο στο Μογκαντήσου, το οποίο γενιάστηκε τον Αύγουστο από την Κάθριν Άστον. Και έχουμε τις ε, τρεις ε, αυτές αποστολές, στρατιωτικές και μη στρατιωτικές, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται. Πώς καταμετράμε τώρα, πώς αποτιμούμε την επιτυχία. Δύσκολο είναι αυτό να το κάνει κανείς με αριθμητικό τρόπο. Αν δούμε όμως τα αποτελέσματα της Αταλάντα, βλέπουμε ότι έχουμε και κάποια ποσοτικά στοιχεία τα οποία είναι ιδιαίτερα θετικά. Νομίζω ότι πέντε μόνο πλοία έπεσαν θύματα πειρατείας, ενώ το 2011 είχαμε 65 και δεν οφείλονται μόνο οι καιρικέ συνθήκες σε κάτι τέτοιο, η επιχείρηση Αταλάντα χρησιμοποιεί όλο και καλύτερα μέσα προστασίας των πλοίων. Σε πάρα πολλά εμπορικά πλοία έχουμε καταφέρει να εγκαταστήσουμε κάποιες στρατιωτικές μονάδες, στρατιώτες που προστατεύουν τα πλοία αυτά σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη. Και για πρώτη φορά στα πλαίσια της αποστολής μας καταφέραμε πραγματικά να βάλουμε κατά της, του κέντρου διοίκησης των πειρατών. Αυτό έγινε το Μάιο. Για πρώτη φορά χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε βία στα πλαίσια της επιχείρησης αυτής. Αν δείτε γενικότερα πάντως την κατάσταση, όντως η κατάσταση στη Σομαλία έχει τροποποιηθεί. Έχει ε, ολοκληρωθεί πλέον η πολιτική μεταβατική φάση της χώρας αυτής. Υπάρχει μια νέα κυβερνητική διοίκηση στη χώρα. Και ήδη Όλες οι μονάδες που έχουμε καταρτήσει από το 2010 έχουν αναλάβει πλέον δράση. Ελέγχουν όλο και μεγαλύτερη γεωγραφική επικράτεια στη χώρα αυτή. Αυτό θέλαμε ακριβώς να πετύχουμε. Αυτό το οποίο χρειάζεται πλέον είναι περισσότερη συμβολή, συνεργασία και πολιτική υποστήριξη για τις επόμενες φάσεις της πολιτικής μετάβασης. Ένα άλλο παράδειγμα που ανέφερε και ο Πρόεδρος είναι η Γεωργία. Έχουμε εκεί μια επιχείρηση εποπτείας μόνο θα μου πείτε, αλλά έχουμε καταφέρει να συμβάλλουμε πολύ σταθεροποιητικά στη χώρα τελευταία χρόνια μέσω αυτής της αποστολή. Και η αποστολή εκεί πέρα έχει ένα πολύ ξεκάθαρο και ορατό ρόλο είναι από τις ε, μόνες αποστολές με έντονη ορατότητα και αναφέρομαι εδώ πέρα στην αποστολή αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία πραγματικά συμβάλλει και αλλάζει επί τόπου τα πράγματα. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Η Κάθριν Άστον θα αναφερθεί στο ζήτημα αυτό όταν θα έρθει να σας μιλήσει λίγο αργότερα σήμερα. η ερώτηση του κυρίου Κέλεμ και συνέχεια θα μιλήσω πολωνικά. Όσον αφορά τη Λιβύη, Όντως εδώ πέρα πρέπει να έχουμε πρόσβαση στους σωστούς ανθρώπους. Θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο, αλλά βλέπουμε ότι τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Δεν καταφέρνουμε να βρούμε τους σωστούς συνομιλητές. Αυτή την εμπειρία είχα και εγώ όταν πήγα νωρίτερα το Φεβρουάριο στη Λιβύη κατά τη διάρκεια της πολιτικής μεταβατικής περίοδου και όλοι οι συνομιλητές με τους οποίους ήρθα σε επαφή εξαφανίστηκαν τελικά από το πολιτικό προσκήνιο μετά από δύο-τρεις μήνες. Είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να εντοπίσουμε κάποιον υπεύθυνο για λήψη αποφάσεων στη Λιβύη δεν καταφέρνουμε ουσιαστικά να στείλουμε κάποιον στη Λιβύη ακριβώ για αυτό το λόγο και για λόγου ασφάλεια επίση. Ξέρετε πόσο ρευστά τα πράγματα στην χώρα αυτή και πρέπει προφανώ εμεί να προστατεύσουμε δεόντω του άντρε και τι γυναίκε που στέλνουμε στη χώρα αυτή. Είπατε ότι χάσαμε μια ευκαιρία. Ξέρουμε όμως ποια είναι η ιστορία που κρύβεται πίσω από το όλο συμβάν. Προφανώς θέλουμε να έχουμε μια πιο φιλόδοξη συμμετοχή στην Λιβύη τα διδάγματα τα οποία έχουμε αποκομίσει είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και για το σχεδιασμό και για το στρατιωτικό δυναμικό που θα έπρεπε να είχαμε στη χώρα αυτή και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πολύ σημαντικό δίδαγμα για το pooling and sharing και για τη νέα δομή που θέλουμε να ακολουθήσουμε στα πλαίσια του pooling and sharing στο μέλλον. Και πώς θα μπορούσε αυτό ακόμα και να συμβάλλει περισσότερο σε έναν καλύτερο εναέριο ανεφοδιασμό καυσίμων. Ξέρετε ότι πριν από ένα χρόνο είχαμε μία ακρόαση για το ζήτημα αυτό και η κατάσταση βέβαια δεν έχει τροποποιηθεί πολύ. Όσον αφορά τώρα τον κώδικα συμπεριφορά, προφανώ εμεί δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πράγματα. Μπορούμε πάντω να βοηθήσουμε στο να βελτιωθούν κάπω τα πράγματα, να ενθαρρύνουμε ουσιαστικά τα κράτη-μέλη να δείξουν μεγαλύτερη διάθεση συνεργασία, να προωθήσουν περισσότερο κάποια συγκεκριμένα σχέδια. Εμεί αυτό το ονομάζουμε mainstreaming θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε pooling and sharing και γενικότερε επενδύσει που έχουν γίνει σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να βελτιώσουμε τη γενικότερη συμβολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο έχει γίνει για παράδειγμα στη Σουηδία, όσον αφορά τώρα την ευελιξία και τι μάχημε μονάδε. Δύο πράγματα εδώ θα μπορούσα να πω. Πρώτον, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πολλές διαφορετικές συνιστώσεις, να χρειαζόμαστε ένα, μια ιατρική συνιστώσα, μια ιατρική μονάδα, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τη χρησιμοποιούμε και τέτοιες ανάγκες έχουμε εντοπίσει στο παρελθόν. Στα πλαίσια συγκεκριμένων επιχειρήσεων χρειαζόμασταν δεσμευμένες ιατρικές μονάδες τις οποίες δεν μπορούσαμε να βρούμε. Μια άλλη ιδέα που ακούστηκε στο παρελθόν και που θα μας απασχολήσει και τις επόμενες εβδομάδες είναι στα πλαίσια συγκεκριμένων μάχημων μονάδων να έχουμε και μη στρατιωτικές συνιστώσεις χωρίς όμως να πρέπει να αλλάξουμε όλη την αντίληψη και τη δομή των ε, στρατιωτικών, των μάχημων μονάδων. Να μπορούμε δηλαδή κάθε φορά να προσθέτουμε και μία μη στρατιωτική συνιστόση, μία ιατρική συνιστόση, όπως σας είπα πριν από λίγο. Κάτι τέτοιο έχουμε δει και στο Αφγανιστάν. Συνεχίζει στα πολωνικά ο μιλητής. Θα αναφερθώ τώρα στην ερώτηση του κυρίου Ζήμκε για τις ομάδε ομάδες μάχης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πολλές φορές οι εμπειρίες που έχουμε είναι ιδιαίτερα οδυνηρές. Εδώ και 7 χρόνια προσπαθήσαμε να δώσουμε μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο ορισμό για τη μάχημη μονάδα χωρίς να έχουμε την απαραίτητη επιτυχία. Ένα ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει πολλές φορές στις συζητήσει των Υπουργών Άμυνας είναι το εξής, να χρησιμοποιήσουμε τις μάχημες μονάδες ως αποθεματικό κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αυτό έχει ακουστεί και την περίπτωση της Βοσνίας για την επιχείρηση που έχουμε εκεί. Έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια μάχημη μονάδα στην Βοσνία, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική όσον αφορά τις α, μάχημες μονάδες. Ακούστηκε λοιπόν η ιδέα να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο μάχημες μονάδες. Ενδεχομένω η προσέγγιση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι κάπως μία ήπια προσέγγιση, πάντο αποτελεί μια θετική αρχή τουλάχιστον. Αναφερθήκατε σε έναν νεαρό Πολωνό, ο οποίο έχασε τη ζωή του στο Μαλί. Θα μπορούσε προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει, αλλά μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε καν προξενική εκπροσώπηση στη χώρα αυτή. Υπήρχαν ορισμένα κράτη-μέλη που είπαν ότι θα πρέπει καταρχά να έχουμε μία προξενική εκπροσώπηση στη χώρα αυτή, πρωτού κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Άλλες ε, χώρες είπαν ότι θα έπρεπε να γίνει μια διαφορετική προσέγγιση, ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν μια διαφορετική προσέγγιση. Την Παρασκευή πάντως ε, θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με συνομιλητές στη χωρα αυτη πρωτου κανουμε οτιδηποτε αλλο Άλλε χώρε ειπαν οτι θα επρεπε να γινει αυτή, βάσει των ε, δομών που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό πάντως και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στη Συρία, να καταφέρουμε να συμβάλλουμε, να βοηθήσουμε τις οργανώσεις που μπορούν να μας υποστηρίξουν στην χώρα αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Bien, merci λοιπόν, ευχαριστώ. Κλείνουμε αυτό το πρώτο τμήμα των ανταλλαγών απόψεων με τον κύριο Ποπόφσκι και τώρα θα περάσουμε στην ετήσια έκθεση για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας που προετοίμασα εγώ ίδιος και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Κατατέθηκαν 198 τροπολογίες και πραγματικά θα πρέπει να συμμολογήσω ότι η πληθώρα αυτών των τροπολογιών περιλαμβάνει πολύ σημαντικές συνεισφορές στο κείμενο και οι περισσότερες από αυτές δεν νομίζω ότι παρουσιάζουν δυσκολίες. Προφανώς ορισμένες ε, τροπολογίες έχουν μια πιο πολιτική εμβέλεια η οποία θα πρέπει να συζητηθεί στο πλαίσιο των πολιτικών ομάδων αλλά νομίζω ότι εν γέννη πέρα από κάποιες ε, γνωστές ε, αντιρρήσεις ή ενστάσεις που ήδη έχουν συζητηθεί σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση, θεωρώ ότι γενικά το πνεύμα αυτής της ε, έκθεσης χάνει της αποδοχής της, των περισσότερων πολιτικών ομάδων και θα μας επιτρέψει να έχουμε επικοδομητικές και γρήγορες συζητήσεις για την έκθεση αυτή. Ε, το χρονοδιάγραμμα είναι αρκετά ε, δύσκολο γιατί ε, προβλέπεται στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου μία ψηφοφορία και μέχρι τότε θα έχουμε τη με τους Σκιώδης και θα υπάρξει μια ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ στις 25 Οκτωβρίου προηγουμένως. Βρίσκομαι βεβαίως στην διάθεση των σκιωδών και των συντονιστών των ομάδων, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και πάλι επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει ε, τίποτα σε αυτές τις 198 ε, τροπολογίες που να συνιστά εμπόδια στην επίτευξη μιας ε, συνεννόησης. Θα, βέβαια θα υπάρξει μεσή πιο προβληματικές τροπολογίες. Ε, έχετε διαβάσει την έκθεση, δεν θα σας ξαναπαρουσιάσω τις βασικές γραμμές περιλαμβάνοντας την έκθεση. Φυσικά ε, υπάρχουν ορισμένες διεκδικήσεις αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επανέρχονται ε, σταθερά. Και θέλουμε να υπάρξει μια θετική απήχηση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, το Γενικό Επιτελείο για παράδειγμα που αποτέλεσε αντικείμενο παθιασμένο συζητήσεων στο επίπεδο του Συμβουλίου χωρίς να ε, καταλήξουν σε κάποια λύση. Αυτά είναι από τα θέματα που η κυρία Άστον και οι υπηρεσίες της εκφράζουν σημαντικές επιφυλάξεις το Κοινοβούλιο πραγματικά δικαιώνει το ρόλο του όταν ε, ίσως είναι υπερβολικά, θέτει υπερβολικά φιλόδοξους στόχους για μια βραχυπρόθεσμη εκπλήρωσή τους. Αλλά πιστεύω ότι παράλληλα αυτά θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ορισμένα πράγματα που δεν εισακούονται άμεσα. Ε, είναι μια πρωτοβουλία υπάρχει η Λευκή Βίβλος που έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίες όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Άμυνα και η οποία θα συμπληρώσει την στρατηγική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συντάχθηκε το 2003 και αναθεωρήθηκε το 2008 και θεωρώ ότι είναι όταν σημαντικό γιατί τελικά στάξει μια εποχή ε, γεωπολιτικών αλλαγών και ήταν σημαντικό οι Ευρωπαίοι να αναθεωρήσουν τις προτεραιότητες στον τομέα της άμυνας και να τις συγκεράσουν μαζί με τους περιορισμούς του προϋπολογισμού. Και όλα αυτά σε σχέση με, τους, με τις εθνικές πολιτικές παραμένουν ο ακρογωνίος ε, λήθος της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ε, υπάρχει και ένα κομμάτι που αφορά μια αναθεώρηση των ε, αποστολών στο πλαίσιο της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Αναφέρετε κι εσείς ότι οι περισσότερες αυτές τις αποστολές έχουν θετικό αντίκτυπο. Ε, Ενδεχομένω μπορούμε να πούμε ότι ίσως δεν ήταν αρκετά σημαντική η εμβέλειά τους. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών όσον αφορά τις αποστολές αυτές και επιφέρουν μια προσθέμενη πολιτική στρατιωτική αξία λες, αυτές. Ε, και βεβαίως ε, επιθυμούμε να μην θυσιάζεται η στρατιωτική, το στρατιωτικό στέλος της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Ε, ιδού εν γέννη τα όσα ήθελα να πω ως εισαγωγική, ως εισαγωγή συγγνώμη, και αναμένω τα δικά σας ε, σχόλια. Και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους συντονιστές και στους ε, σκιώδες για να γίνει η συζήτηση. Ωραία λοιπόν. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ ευγνώμων για αυτό το υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών, γιατί δεν είμαστε πάντοτε σε θέση να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών από την πλευρά της Realpolitik, αλλά πάντοτε αποτελεί μια πηγή υψηλής έμπνευσης και αναφέρατε τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τα επιτελεία των ε, επιχειρήσεων. Είναι ένα θέμα που το συζητούμε επί μήνες. Εξετάσαμε τις ε, διάφορες εναλλακτικές ε, προτάσεις, αλλά μία ρεαλιστική λύση ενεργοποίησης του επιχειρησιακού στρατηγίου έχει γίνει ε, ούτως ώστε να συνδράμει τις επιχειρήσεις και αποστολές στο κέρας της ε, Αφρικής. Και θέλουμε να είμαστε πραγματιστές και να συνεχίσουμε ε, σε αυτή την πορεία. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια στην έκθεση, χωρίς να είμαι εγώ θα εξαντλήσω όλα τα θέματα. Καταρχήν αναφέρεται σωστά στο το στρατηγικό πλαίσιο και έτσι κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια νέα στρατηγική ασφάλειας. Ε, διεξάγεται εδώ και πολύ καιρό και οι ευρωπαϊκές χώρες έθεσαν κάποιες νέες συνιστώσεις μιας νέας ε, στρατηγικής ασφάλειας, άλλες ήταν πιο επιφυλακτικές. Ε, κατ' εμέ σημαντικός είναι ένας στρατηγικός προβληματισμός ως προς τα πού θέλουμε να κινηθούμε. Τώρα το πλαίσιο αλλάζει λόγω της ε, αναμενόμενης ε, συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και νομίζω ότι αυτή είναι μια χρυσή ευκαιρία για μας να κάνουμε μια περιεκτική και εισβάθα συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, πέρα από τις τρέχουσες υποθέσεις. Ε, ε, και ε, βεβαίως η συζήτηση αυτή κάπως έχει ανοίξει ε, ότι ε, να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό στην Ευρώπη το οποίο θα πρέπει να αξιοποιήσουμε. Δεν παίρνουμε κάποια ε, τελική θέση. Είναι μια σύντηση μεταξύ κυβερνήσεων και ενεχομένων πλευρών. Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σε αυτό το πλαίσιο. Και βεβαίως σημειώνουμε ε, το όσα είπατε για μια λευκή βίβλο. Και δεν λέω ότι η συζήτηση με τους επακεφαλείς των κυβερνήσεων θα υποκαταστήσει την ανάγκη της λευκής βίβλου. Αλλά πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση και θα δούμε τι θα συμβεί στις ενδιάμεσες φάσεις αυτής της συζήτησης, την οποία ήδη ε, ε, και έχουμε ήδη, έχει ήδη ξεκινήσει μια συνάντηση των υπουργών, θα γίνει ήδη μια συνάντηση των υπουργών άμυνα τον Νοέμβριο. Τώρα, όσον αφορά μια τέτοιου είδους ε, προσέγγιση, με τον Άιδος στις θρησκείας στη Βρυξέλλες, γιατί όλοι αναποθέτουν εκεί τις ελπίδες τους. Και αυτά, σας περιέγραψα το τι γίνεται στις επιχειρήσεις των χεράς της Αφρικής, πραγματικά πήγαν καλά. Αλλά θα ήθελα να είμαι απολύτως ξεκάθαρος προς το θέμα αυτό. Μια περιεκτική προσέγγιση ε, δεν είναι ένας τρόπος να αμβλύνουμε τη στρατιωτική διάσφαλιστικό στέλος της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Ε, δεν ε, είναι μια υποκατάστασή αλλά είναι το κοινό πλαίσιο εντό του οποίου ε, αξιοποιούμε τα εργαλεία πολιτικής αλλά και στρατιωτικής διαχείρισης των κρίσεων όπου έχουμε ένα περιεκτικό πλαίσιο όπως το Σαχέλ ή το κέρας Αφρικής, ε, η το κερες πολιτική ασφάλειας άμυνας και άμυνας αναπτύσσεται εκεί γιατί ξεκινήσαμε με την ε, στατική επιχείρηση της ε, Αταλάντης και μετά προσθέσαμε στρατηγικό πλαίσιο. Στα χέρια έγινε το αντίστροφο. Ε, καταρχήν πήραμε μια απόφαση για το στρατηγικό πλαίσιο και στη συνέχεια το συμπληρώσαμε με διάφορες δράσεις. και η τελευταία είναι η UCAP στο Νίγηρα και η νέα αποστολή που αρχίσαμε να συζητούμε στο Μαλί. Άρα λοιπόν πρόκειται για ουσιαστικά πράγματα που πραγματικά κάνουν τη διαφορά εδώ. Ε, δεν ξέρω αν έκανα συγκεκριμένα σχόλια για τις επιχειρήσεις εδώ μπορώ να επανέλθω εάν θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο. Εν γέννη, ε, οι σκέψεις σας μας βοηθούν βεβαίως στην διαμόρφωση αυτής της συζήτησης ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τη συζήτηση που θα γίνει. Ίσως θα ήθελα να κάνω τρία πιο ξεκάθαρα σχόλια για την κυβερνοασφάλεια και τις νέες τάσεις. Για τις νέες απειλές, συγγνώμη. Είπα ότι εκπρόσωπος πήγε την περασμένη εβδομάδα στην διάσκεψη για την κυβερνοασφάλεια ε, και περιέγραψε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια νέα ε, ανακοίνωση που θα εκδοθεί και το θέμα αυτό της κυβερνοασφάλειας, ε, κοινή ανακοίνωση. Και μετά από αυτή τη συνάντηση θα πάω στο Συμβούλιο για να συζητήσουμε τι γίνεται όσον αφορά το θέμα της κυβερνοασφάλειας στο επίπεδο των χωρών μελών. Ένα άλλο στρατηγικό θέμα το οποίο θα μπορούσε να μας βοηθήσει να ορίσουμε επακριβώς μια κοινή γραμμή, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, προδιαγραφές υπεύθυνη συμπεριφορά στον κυβερνοχώρο, που είναι κάτι θεμελιώδες, γιατί πρόκειται για ένα χώρο ο οποίος δεν είναι αρκετά ρυθμισμένος, αντίθετα θα έλεγα. Επίσης, όσον αφορά το διάστημα, αναφερθήκατε στο θέμα του διαστήματος στην έκθεσή σας. Ε, πράγματι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ο λεγόμενος ε, Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας ε, για το διάστημα το οποίο ξεκινήσαμε διάφορους μας στον κόσμο με τις ΗΠΑ για παράδειγμα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε μία συμφωνία. Δεν έχουμε ακόμα ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα γιατί θα πρέπει προηγουμένως να πείσουμε κάποιους άλλους εταίρους μας αλλά πραγματικά πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα το οποίο ε, παρακολουθώ εκ του σύνεγγυς εγώ ο ίδιος εκ μέρους της είπα της εκπροσώπου. Και τέλος ένα ειδικό θέμα το οποίο αναφέρατε στην έκθεσή σας και πάλι κάτι το οποίο εξετάζουμε επίση η ενίσχυση της ε, εμπειρογνωμοσύνης στις αποστολές των Ηνωμένων Εθνών. Σε πολλές από αυτές τις αντιπροσωπείες μας συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε έναν αξιωματούχο, ένα σύνδεσμο στην ε, Πούτζα και νομίζω ότι είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο γιατί έχει την εντολή να απευθύνει συμβουλές στον τρόπο που ε, δεσμευόμαστε με την ΙΚΟΑΣ, την Οικονομική Κοινότητα Δικαιωτικοαφρικών ε, Κρατών και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα μαζί τους. Μετά από αυτή τη συνάντηση, όπως είπα, θα πάω στο Συμβούλιο και το δεύτερο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τις χώρες μέλη είναι αυτό ακριβώς το θέμα της εμπεριγνωμοσύνης και θα θέλαμε να περιγράψουμε τις, τους δικούς μας προβληματισμούς και υπάρχει μεγάλη ζήτηση εδώ. Άρα το θέμα αυτό είναι πολύ κέριο γιατί και οι ίδιοι επικεφαλείς των αντιπροσωπιών θέλουν να έχουν μια εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας, ιδιαίτερα σε εκείνες τις χώρες όπου έχουμε αναλάβει δράση και έχουμε κάποιες ε, επιχειρήσεις και αποστολές, να υπάρχει κάποιος ο οποίος να απευθύνει ειδικέ ε, συστάσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Για το τελευταίο αυτό σημείο συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και αυτό άλλωστε αποτέλεσε και αίτημα των επικεφαλής των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιοχές εκείνες του κόσμου που δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αποστολών κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, αλλά και με τις χώρες εκείνες που θα μπορούσαμε να συνάψουμε εταιρικέ σχέσεις, με τρίτες χώρες δηλαδή, με χώρες οι οποίες επιθυμούν όλο και περισσότερο να δούνε αποστολές κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, η Κίνα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για διάφορες αποστολές καταπολέμησης της πειρατείας. Ο αντιπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πεκίνο μας είπε ότι οι ε, εκεί υπεύθυνοι θα θέλανε να είχαν και τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να καταφέρουν να συμπληρώσουν τη δική τους δράση. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον σκιώδη εισηγητή μας, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη διότι ήρθαμε μια μικρή καθυστέρηση. Είχατε ήδη κάνει την εισαγωγική σας παρέμβαση ως εισηγητής για το ζήτημα αυτό. Για το σχέδιο έκθεσης για την εφαρμογή της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Ξέρετε όμως πώς είναι οι κοινοβουλευτικές εργασίες. Έπρεπε να ψηφίσω στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ε, ε, μία έκθεση στην οποία ήμουν ασκιώδης συζητητή και ε, μόλις τελείωσε ήρθα εδώ στη συζήτηση που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό θέμα που έχουμε για όλη τη θητεία μας. και σε γενικές γραμμές ε, συμφωνώ με τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις ε, ε, της εκθέσης του κυρίου Νταζάν και πέραν αυτού όμως έχουμε παρουσιάσει και κάποιες τροπολογίες για κάποια θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα ή μας απασχολούν ιδιαίτερα. Ε, στόχος μας είναι να ενισχύσουμε και να επισημάνουμε την αναφορά στον αποτελεσματικό ε, συνολικό ε, αντιμετώπιση των θεμάτων είναι και κάτι το οποίο επισημάναμε την τελευταία δεκαετία και θέλουμε να το ενισχύσουμε ιδιαίτερα. Είναι πολύ σημαντικό ε, και σημαίνει κατά βάση σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ε, στα όσα προτάνουν τα ενωμένα Έθνη είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναφέρεται συνεχώς αυτό. Επίσης ε, θέλουμε να υπάρχει και συγκεκριμένη μνήμα στην αρχή της ευθύνης ε, προστασίας. Είναι κάτι σχετικά νέο από πλευράς Ενωμένων Εθνών και προέκυψε λόγω της ε, διάδοσης των συγκρούσεων και επειδή υπήρχε αδράνεια από πλευράς διεθνούς κοινότητας ή ε, πολύ ελλειπής ε, δράση, διότι δεν υπήρχε νομική κάλυψη και αυτό σημαίνει ότι ολόκληροι λαοί και στο παρελθόν και τώρα καταπιέζονται από τους ηθήνοντες ή από τους τυράννους τους. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας καταδεικνύει ότι υπάρχουν δυνατότητες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να δράσει ως παγκόσμιος παράγοντας και μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα μέσα της υπέρ αυτής της ε, κοινή πολιτικής ασφαλείας και στρατιωτικές και πολιτικές δυνάμεις, ε, χρηματοοικονομική στήριξη. Ε, όλα αυτά σημαίνει ότι υπάρχουν δυνατότητα για να θέσει όρους, για να επηρεάσει και να έχει και μια θετική επιρροή και να μπορέσει να πιέσει στο παγκόσμιο πλαίσιο στο οποίο κινείται η Ευρώπη. Και επίσης ε, αυτή η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας είναι σημαντική και για την ε, διατλαντική μας συμμαχία και πρέπει να μπορέσει να διασφαλίσει και τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Μια Ευρώπη ε, που έχει πάρα πολλές δυνατότητες ωφελεί ιδιαίτερα το ΝΑΤΟ και πολλές φορές εδώ στο Κοινοβούλιο έχουν συζητηθεί οι σχέσεις ε, και οι, δυνα... οι πιθανές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Πέραν αυτού όμως εγώ βλέπω και μια απαραίτητη συμπληρωματικότητα και αυτό ε, διαπιστώνεται καθημερινά. Είναι περισσότερη αυτή η συμπληρωματική πτυχή και όχι η... η ε, διαφιλονικίες και διαμάχες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Θέλουμε να βελτιώσουμε λοιπόν ε, την ε, ε επιχειρησιακές δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμενας και να είναι συντονιστής ε, και να καθορίζει παρα, εκ παραλίλου προγράμματα τα οποία θα δρουν με τα κράτη-μέλη. Πρόκειται για μόνιμο στόχο του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουμε να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις και να μην τριπλασιάζονται ή να πολλαπλασιάζονται δαπάνε ε, για πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει κάλλιστα κάποιο άλλο τομέα, Το να γίνονται πράγματα από κοινού είναι μόνιμο στόχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τέλο έχουμε προσθέσει και κάποιε τροπολογίε που αφορούν ε, τη μη διάδοση των όπλων και τον αφοπλισμό ε, τις ε, δυνατότητες που έχουν οι ασιατικές χώρες και η Κίνα για την παγκόσμια ασφάλεια. Νομίζω ότι λόγω απόστασης ε, δεν δίνουμε τη δέουσα προσοχή στον τρόπο με τον οποίο εξοπλίζεται η Ασία, ε, κυρίως η Κίνα, και το οποίο θα μπορούσε ίσως να επηρεάσει την παγκόσμια ασφάλεια. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές. Όσον αφορά τώρα τη στρατηγική ασφαλείας, την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας, Έχω την εντύπωση ότι η ύπατη εκπρόσωπος και η υπηρεσία της ε, δεν είναι υπέρμαχη αυτή τη στιγμή ε, της ανανέωσης μιας στρατηγικής η οποία εγκρίθηκε το 2008 και ακόμα είναι εξελίξει σε κάποιες πτυχές της. Ο εισηγητής όμως ε, είναι υπέρμαχος αυτή τη δυνατότητα. θα το συζητήσουμε στις συνεδρίες με τους συντονιστέ την επόμενη εβδομάδα και θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε ίσως σε κάποιο συμβιβασμό για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup, Madame <coughs> ε, Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, εδώ πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα και από τη δική μας πλευρά της ε, ΓΚΟΕ δεν μπορώ να επισέλθω σε όλες τις πτυχές αυτής της έκθεσης, γι' αυτό θα ήθελα εδώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις γενικής φύσεως. Από τη δική μας σκοπιά και κατά τη δική μου προσωπική άποψη η έκθεση αυτή ακολουθεί και αυτό ισχύει και για την συζήτηση που κάναμε προηγουμένως ακολουθεί ε, ένα τραγικό γνώμονα της ε, ανθρώπινης ε, δράσης όπως όταν ε, για παράδειγμα οι γονείς που δέρνουν τα παιδιά τους για να είναι καλύτερα στο σχολείο, είναι καλύτεροι μαθητές, αλλά ε, τα παιδιά γίνονται ακόμα χειρότεροι μαθητές, τα οι γονείς τα δέρνουν όλο και πιο πολύ, αυτά χειροτερεύουν όλο και πιο πολύ, τα δέρνουν όλο και πιο πολύ κλπ. Δηλαδή είναι μια ε, περαιτέρω ανάπτυξη εσφαλμένης πρακτικής αυτός ο γνώμονας της ανθρώπινης πράξης. Ο κύριος Ντανζόν γράφει στην έκθεσή του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται διεθνώς ε, να δράσει ως ε, πολιτικός παράγων προκειμένου να εξασφαλίσει και να προωθήσει τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και να προστατεύσει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ολόκληρο τον κόσμο και να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών της. Προηγουμένως ε, τέθηκαν κάποιες ερωτήσεις κατά πόσο πράγματι μέσω όλων αυτών των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ ή των κοινών ε, αποστολών να έχει ε, βελτιωθεί πράγματι η κατάσταση ε, στον κόσμο, να ε, έχει πάψει καταπίεση, καταστολή, έχουν πραγματικά προστατευτεί αποτελεσματικά τα συμφέροντα των πολιτών. Θα πρέπει να διαρωτηθούμε ποια είναι η κατάσταση των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, ποια είναι η κατάσταση των ανθρώπων σε πολλέ άλλε χώρε του κόσμου. Σε αυτές τις ερωτήσεις δίδει ο εισηγητής την απάντηση που υπακούει ακριβώς σε αυτό το βασικό γνώμονα ε, που σας περιέγραψα. Ε, απαιτούνται πιο σκληρές ε, παρεμβάσεις και αποστολές και επιχειρήσεις σε περισσότερα μέρη του κόσμου. Κατά την άποψή μου αυτή είναι μια πραγματικά τραγική γραμμή που ακολουθούμε. Ε, και θα ήθελα κλείνοντας να αναφερθώ στον παράγοντα του κόστους, γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην Ευρώπη όπου ε, η κοινωνική περίθαλψη των ανθρώπων σε πάρα πολλές ε, χώρες έχει καταστραφεί σχεδόν. Ε, για παράδειγμα στην Ελλάδα έχει καταρρεύσει το σύστημα υγείας. Και στην έκθεση αυτή επικρίνεται το γεγονός ότι περικόπτονται κάποιες δαπάνες. Από 288 δις το 2010 ε, ε, έγιναν κάποιες περικοπές ε, το 11 και αυτό επικρίνεται και διατυπώνεται το αίτημα να προωθηθεί η εξοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σημαντικότερο παράγοντα για την ειρήνευση κλπ. Εγώ νομίζω ότι η πιστική είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο εφόσον επιτυγχάνει να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων στις χώρες όπου παρεμβαίνει με πολιτικό τρόπο ακριβώς την, ε, τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών και όχι του πολιτοστρατιωτικού ε, συμπλέγματος, αν θέλετε, του πολιτοστρατιωτικού μπλοκ ε, στην Ευρώπη. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Η κυρία Κοπά έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι τον Πρόεδρό μας για την έκθεσή του και να σχολιάσω εν συντομία τις τροπολογίες. Η πρώτη μου γενική παρατήρηση αφορά την, τύση, την τάση να συγχαίουμε τις φιλοδοξίες μας με την πραγματικότητα των δυνατοτήτων μας και όπως αναφέρθηκε και στην έκθεση Λίζια και επιβεβαιώνει και η έκθεση Ντανζάν, τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν δύσκολους καιρούς και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουν περικοπές στις αμυντικές τους δαπάνες. Επομένως, θα πρέπει να βρούμε τρόπους να διασφαλίσουμε τις απαραίτητες δυνατότητές μας, να διασφαλίσουμε ότι είναι ασφαλείς οι ευρωπαϊκοί πολίτες και να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στην διατήρηση της ειρήνης και την ενίσχυση της διεθνούς ασφαλείας στα πλαίσια της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή είναι μια απαραίτητη ρεαλιστική προσέγγιση δεδομένων των συνθήκων ε, διαπιστώνω όμως ότι κάποιοι από εμά συγχαίουν ε, το γεγονός αυτό με μια απόπειρα να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια υπερδύναμη. Και στις τροπολογίες διαπιστώνω ότι υπάρχει ε, μία αιμονή σύγκρισης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων αναδυόμενων δυνάμεων και ξεχνούν ποιος είναι ο στόχος της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Ακόμα και αν θα θέλουμε ε, να γίνει υπερδύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι ούτε υπερδύναμη ούτε υπερκράτος και επομένως δεν μπορεί να αντιμάχεται τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το ίδιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, όπως ε, εγγράφεται στη συνθήκη, είναι ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιούμε με σοφροσύνη η κοινή πολιτική άμυνας, ασφάλειας και άμυνας είναι λίγο παραπάνω από τα λεγόμενα καθήκοντα της Πετρούπολης και θα πρέπει απλώς να βοηθά στις στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές. Όσον αφορά τις στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές, έχω ήδη ή κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων ότι δεν θα πρέπει να έχουμε απόλυτα αρνητικό τόνο στην έκθεση. Συμφωνώ όμως ότι θα πρέπει να τηλήσουμε διδάγματα από το παρελθόν και ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει επίσης να κάνουμε και αξιολόγηση των ενεξελίξεων αποστολών με στόχο να καταργήσουμε αυτές οι οποίες ίσως είναι πλέον ε, περιτές. Στα Δυτικά Βαλχάνια, για παράδειγμα, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα προβλήματα ναι με ενεμένουν ναι αλλά δεν αφορούν μόνο την διάσταση της ασφάλειας και θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη σημασία στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Οι δύο τελευταίες παρατηρήσεις μου αφορούν τις επιπτώσεις ε, της ε, κρίσης ε, στην ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση και το pooling and sharing. Αν συνεχιστεί η κρίση, η βιομηχανική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συρρυκνωθεί, θα υπάρχουν απώλειες θέσεις εργασίας και θα υπάρχει μεγάλης κλίμακας μετανάστευσης ανθρώπων με υψηλές δεξιότητες και γνώσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προάγουμε ευρωπαϊκές συνέργειες και να είμαστε υπέρ ενός ευρωπαϊκού προγράμματος προγράμματος το οποίο θα είναι ανοιχτό ως ε, αρχή σε όλα τα κράτη-μέλη προς συμμετοχή. Με άλλα λόγια, δεν πιστεύω τόσο πολύ στις διμερείς πρωτοβουλίες και πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει και σε νέο ανταγωνισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο αφορά και τις ε, διμερείς συνεργασίες σε θέματα pooling and sharing. Θα πρέπει λοιπόν να εκφράσουμε την πλήρη στήριξή μας για ένα pooling and sharing το οποίο θα περιλαμβάνει τους πάντες και να ε, επιδοκιμάσουμε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας για να υπάρχει ένα κώδικας διοντολογία για το pooling and sharing, το οποίο είναι κάτι το οποίο εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα από του ε, Υπουργού Άμυνα Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άτυπη σύνοδό του, ε, την οποία φιλοξώνησε η Κυπριακή Προεδρία. Και με τη συμφωνία του εισηγητή μας και όλων σας θα μπορούσαμε να έχουμε και μια προφορική ε, τροπολογία για να λάβουμε υπόψη και τις τελευταίες αυτές εξελίξεις. Ευχαριστώ. Λίγα λεπτά έχουμε ακόμα στην ε, διάθεσή μας για να ακούσουμε και άλλες ε, παρατηρήσεις. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά γιατί πραγματικά οι περισσότερες τροπολογίες είναι ιδιαίτερα επικοδομητικές και θα τις διατηρήσουμε πιστεύω. Βλέπω ότι εμένεται ιδιαίτερα σε αυτά που είπε και ο κύριος Γιαννιές και ορισμένοι συναδελφοί του, δηλαδή να γίνεται μία αναφορά στον πολύπλευρο χαρακτήρα, στο ότι θα πρέπει πραγματικά να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, τους πολίτες, τους κατοίκους, τις περιοχές που επεμβαίνουμε και ότι θα πρέπει να ενσωματώσουμε τη διάσταση αυτή πλήρως Σαφώς θα μπορούσαμε να εμένουμε στην διάσταση αυτή, αλλά νομίζω ότι άλλωστε η ε, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ούτως ή άλλως εμένουν στο ζήτημα αυτό, ούτως ή άλλως εμπεριέχουν αυτή τη συνιστόσα. Θα μπορούσαμε πάντως να δώσουμε μεγαλύτερη προβολή, αν θέλετε, σε αυτή τη διάσταση. Θα ήθελα να επιθυμίσω επίσης όλους τους συναδέλφους ότι εξετάζουμε αυτή τη στιγμή μια συγκεκριμένη έκθεση που έχει να κάνει με την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνας και θα πρέπει να δώσουμε αξιοπιστία ακριβώ στη διάσταση αυτή, τη ασφάλεια και τη Άμυνα. Κάποιε πιο γενικέ παρατηρήσει μπορούν να συμπεριληφθούν σαφώ, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην έκθεση για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια του κ. Μπρόκα. Δεν έχω να κάνω άλλες ειδικέ παρατηρήσεις. Ορισμένοι συνάδελφοι ανεξαρτήτως πολιτικής ομάδας θέλησαν να συμπεριλάβουν την ΕΜΠΑ Μολδαβή, την επιχείρηση αυτή στη Μολδαβία, στην έκθεση. Η επιχείρηση αυτή όμως δεν είναι επιχείρηση της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και αυτό το λόγο δεν την συμπεριέλαβα ανεξάρτητα από το πόσο καλή ή όχι είναι η αποστολή αυτή, αποτελεί αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να λάβω υπόψη μου τις σχετικές τροπολογίες που θέλαν την ένταξη της αποστολής αυτής. Ορισμένες πολιτικές ομάδες κάνανε κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο κέρας Αφρικής. Νομίζω, νομίζω ότι εκτενώς καλύψαμε το ζήτημα αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μιλήσουμε περισσότερο στο στάδιο αυτό. Οι σκιώδεις ηγητές θα συνεδριάσουν στις 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και μία ακόμα συνεδρίαση στο Στρασίκο 3 Οκτωβρίου. Και μέχρι τότε προφανώς θα είμαστε σε στενή επαφή για να καταφέρουμε να ενσωματώσουμε όλες αυτές τις τροπολογίες. Εν γέννη πάντως πιστεύω ότι δεν θα συναντήσουμε σημαντικές δυσκολίες. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ, ευχαριστώ και τον κύριο Ποπόφσκι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε να μας δείτε. Νομίζω ότι η τακτική ενημέρωση ε, είναι πάρα πολύ σημαντική για μας όσον αφορά τα ζητήματα την οποίων άπτεται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα όσον αφορά και την αποστολή στον Νίγηρα για να δούμε τελικά πόσο αποτελεσματική είναι. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά πολύ και περιμένουμε και τον κύριο Μπρόκ. Κύριο Μπρόκ, έχει το λόγο. Ναι, ναι. Σα υπενθυμίζω λοιπόν ότι περιμένουμε την ύπατη εκπρόσωπο και ότι θα γίνει και κλεισμένο το θυρών η συνεδρίαση. Μόνο τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το προσωπικό των πολιτικών ομάδων, καθώς επίσης και των επιτροπών και σχετικών υποεπιτροπών και τα μέλη των γενικών διευθύνσεων αρμόδων για τα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η άλλη θα πρέπει να αποχωρήσετε από την αίθουσα, παρακαλώ.